Good afternoon, colleagues, and we begin with point 20. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Ξεκινούμε σημείο 20. Παρασίωση, παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Ανακοίνωση για τη διατήρηση και την ένωση του Σέγγεν. Υιοθέτησε το Σεπτέμβριο η Επιτροπή το πακέτο μια ανακοίνωση για τη διαφύλαξη του κεκτημένου, σύσταση για την εφαρμογή του κανονισμού για τα σύνορα, προστασία των ιστορικών σύνορων του χώρου Σέγγεν και νομοθετική πρόταση που τροποποιεί τις διατάξεις. Πρόκειται για τη σύσταση παριθμών 399. Και θα παρακαλέσω τον κύριο τεκόιστα τώρα να μας κάνει την παρουσίαση αυτής της δέσμης και να απαντήσει μετά στις ερωτήσεις. Κύριε Τεκούστα, σας ακούμε και μετά θα ακούσουμε τους βουλευτές. Οι συγκητές πρώτα και μέλη της Επιτροπής. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο Επίτροπος χθες ε, έλαβε αποφάσεις που με διευκολύνουν στη σημερινή μου παρουσίαση για το σημείο 9 της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση και την Υλοποίησή του παρουσίασε σύντομα και την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση του Σέγγεν, διατήρηση και ενίσχυση του Σέγγεν. Κύριο συμπέρασμα ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις Σέγγεν για την προσωρινή επαναφορά των ε, ελέγχων στα σύνορα τα ιστορικά σύνορα, σύνορα Σέγγεν και παρουσίασε ο Επίτροπος τα κύρια σημεία και βέβαια πάνω σε αυτά θα αναπτύξω κι εγώ. Πριν όμως περάσω αυτήν την νομοθετική πρόταση, επιτρέψτε μου σύντομα να υπενθυμίσω την εξέλιξη στη ρήτρα διασφάλισης του Σέγγεν, δηλαδή τη διατάξη για την προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει στην απόδειξη ότι είναι μια λογική περαιτέρω εξέλιξη η εξέλιξη αυτή στην πορεία του Σέγγεν και σε σχέση με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο χρόνια τα κράτη Σέγγεν. Σύμβαση Σέγγεν λοιπόν 1990. Άρθρο 2. Για πρώτη φορά ενσωματώνεται η ρήτρα διασφάλισης που έχει την εξής διατύπωση. Αφού προσδιορίστηκε η αρχή της άρσης των εσωτερικών ελέγχων στα σύνορα, ε, λέει λοιπόν, εάν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, ένα συμβαλόμενο μέρος, κατόπιν διαβουλεύσουν με άλλα συμβαλόμενα μέρη, μπορεί για περιορισμένη χρονική περίοδο να άρει να επαναφέρει μάλλον τους εσωτερικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και αυτό μπορεί να δει και παράταση. Άρα η προσωρινή επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα υπήρχε χωρίς όμως μέγιστη περίοδο διάρκειας των ελέγχων αυτών και προβλέπει διαβουλεύσεις. Αυτό ήταν όλο. Επιβίωσε επί 12 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο Σέγγεν με αυτή την ε, πολύ απλή ρήτρα διασφάλιση, γιατί τα περισσότερα κράτη που την εφάρμοζαν, την επικαλούνταν, την επικαλούνταν για μια-δύο μέρε ή εβδομάδε και αυτόν όλο. Ένα κράτο μέλο μόνο ζήτησε και εφάρμοσε την επαναφορά για αρκετά χρόνια, η εβδομαδε και αυτον ολο ενα κρατο μονο ζητησε και εφαρμοσε την επαναφορα για λόγους σχετικούς με την πολιτική, την ήπια πολιτική για τα ναρκωτικά της, ε, των κατοχωρών. Επαρέφερε λοιπόν η Γαλλία αυτούς τους, συνό, ελέγχους στα σύνορα με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Αλλά δεν φτάσαμε ποτέ στις αποφάσεις αυτές που είδαμε από τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια που για μεγαλύτερη χρονική περίοδο επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους. Το καθεστώς αυτό λοιπόν το 2006 αλλάζει με τον κώδικα, τον συνοριακό κώδικα του Σέγγεν και τη θέσπισή του, που περνάει το διακυβερνητικό εκεί και εκτιμένο του Σέγγεν για του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, διαφυλάσσοντας και τη ρήτρα διασφάλισης, αλλά ταυτόχρονα μιλάει όχι μόνο για κοινοποίηση στα κράτη-μέλη, αλλά και για κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δηλαδή το θεσπικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούσε από την ενσωμάτωσή του στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Σέγγεν. Προσωρινή μόνο επαναφορά των συνόρων ήταν τον ελέγχο στα σύνορα ήταν δυνατή, χωρίς όμως προσδορισμό μέγιστης χρονική περίοδου. Το 2013 και όσοι ήταν μέλη της ΛΥΜΠΕ ήδη τότε θα θυμούνται, υπό το τίτλο Διακυβέρνηση Σέγγεν, όπου παραδείγματι περιλαμβανόταν και ο μηχανισμός αξιολόγησης Σέγγεν, έρχεται μια ουσιαστική τροποποίηση του πεδίου σε σχέση με την διασφαλιστική ρήτρα πολλές νέες διαδικασίες. Η στοιχεία Τμήματα διαδικασιών εισάγονται και για πρώτη φορά επιβάλλεται ανώτατο χρονικό όριο εξάμεινο για την προσωρινή επαναφορά εσωτερικών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Γιατί εξάμεινο. Θα μπορούσαν να ήταν και τρει και εννέα ή δώδεκα οι μήνες. Το εξάμεινο επιλέγει γιατί θεωρήθηκε ότι μπορεί να καλύψει κάθε περίπτωση από αυτές που είχαν μέχρι τότε εμφανιστεί για την επαναφορά των ελέγχων στα ιστορικά σύνορα. Αλλά, άρα απόλυτη αλήθεια ή απόλυτα βάσιμος λόγος για τον οποίο ορίστηκαν αυτοί οι έξι μήνες δεν υπήρξε, αλλά με αυτούς, σε αυτούς έχουμε μείνει στο κώδικα Σέγγεν. Υπήρχε και η δυνατότητα της παράτασης των ιστορικών ελέγχων για δύο χρόνια μόνο υπό το άρθρο 29, το οποίο όμως δεν είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Και τώρα, η Επιτροπή έρχεται με μια άλλη αλλαγή, η πρόταση αλλαγή καλύτερα, της ασφαλιστικής ρήτρας, ιδιαίτερος για να ε, εξασφαλίσει τη δυνατότητα για μια μακρύτερη χρονική περίοδο να να επαναφέρονται οι έλεγχοι στα σωστικά σύνορα. Με την πρότασή της αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Σέγγεν στις ε, προκλήσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα στην ορθή διαχείριση των εξωτερικών ε, ελέγχων ε, συνόρων, την, τις κινήσεις παράνομων μεταναστών, αλλά βέβαια και την τρομοκρατική απειλή. Πρόκειται για προβλήματα που χρονίζουν και φάνηκε ότι οι έξι μήνες ως μέγιστη χρονική περίοδος δεν θα αρκούσαν. Για τις δευτερογενείς κινήσεις που προκύπτουν από ανεπάρκεια στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, η Επιτροπή επεκτείνει και τη διαδικασία του άρθρου 29 με τις συστάσεις που υποβάλλει στο Συμβούλιο, ζητώντας από τα κράτη-μέλη την παράταση με βάση τις συνθήκες και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον κώδικα των συνόρων. Τι κάνει τώρα η Επιτροπή. Προσαρμόζει για άλλη μια φορά, προτείνει την προσαρμογή των ισχυουσών διατάξεων προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα Σέγγεν. Λαμβανωμένων υπόψη, λαμβανωμένων υπόψη όχι μόνο των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη, αλλά και των αντιρρήσεων και επιφυλάξεων που έχουν εκφράσει κάποια κράτη-μέλη που υπέστησαν τις συνέπειες της επανεισαγωγής των ελέγχων στα ιστορικά σύνορα από όμορα κράτη-μέλη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε την πρότασή μας, δηλαδή να βρούμε μια σωστή ισορροπία που θα μας επιτρέπει και να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή περίοδο ε, επιτρεπομένων ελέγχων στα ιστορικά σύνορα για λόγους τρομοκρατίας ή άλλων κινδύνων, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας ότι θα διαταραχθεί ως το δυνατόν λιγότερο η δυνατότητα ιστορικής διακίνησης και ότι θα ενημερώνονται σε όσο δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας τα κράτη-μέλη. Παράταση λοιπόν από τους έξι μήνες στον ένα χρόνο της συνήθους μέγιστης περίοδου κατά την οποία μπορεί να επανεισαχθούν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα. Και αυτό αντισταθμίζεται με μια σειρά από εγγύησεις, επί παραδείγματι, τα στοιχεία της κοινοποίηση. Αυτά ενισχύονται. Με βάση την πρόταση της Επιτροπής πριν από την κοινοποίηση της επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, Πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τα όμορα και συμφωνία πρώτερη για μέτρα συνεργασίας που θα μπορούσαν να αναλυφθούν. Η Επιτροπή έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας πληροφοριών για τη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη-μέλη. Καινοτομία σημαντική επίσης είναι ότι απαιτείται και αξιολόγηση κινδύνου εκτίμηση κινδύνου που θα δείχνει για πόσο διάστημα εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η απειλή, σαφή ορισμό των ε, τμήματων των εσωτερικών συνόλων που μπορεί να επηρεάσει αυτή η απειλή ή οι απειλές που θέλουμε να αποτρέψουμε και επίσης σαφή απόδειξη του γεγονότος ότι η προσωρινή επαναφορά των ε, ελέγχων στα ιστορικά σύνορα είναι η προσωρινη επαναφορα των ελεγχων στα εσωτερικα λύση. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήταν καλό να αναφέρουμε είναι ότι όταν ένα κρατός μέλος ξεπερνά το εξάμεινο για τους ελέγχους στα ιστορικά σύνορα υπάρχει και η υποχρέωση για χορήγηση πληροφοριών για το πόσο μπόρεσαν ουσιαστικά να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ε, κινδύνων αυτή η έλεγχη. Δηλαδή, και δεν είναι πλέον τυπικό στοιχείο της κοινοποίηση, πρέπει να εξηγήσει το κράτος μέλος ε, τι έχει μπορέσει να κάνει καλύτερα, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Επιτροπή, όταν ένα κράτος μέλος ξεπερνά το εξάμεινο για τους ελέγχους στα ιστορικά σύνορα, η Επιτροπή πρέπει να γνωμοδοτήσει. Με τις ισχύουσες διατάξεις η Επιτροπή δύναται να εκδώσει γνώμη και οφείλει να το πράξει εάν έχει αμφιβολίες ως προς την αναλογικότητα ή την αναγκαιότητα των μέτρων. Από τη στιγμή που ένα κρατός μέλος ξεπερνά το εξάμεινο, η Επιτροπή υποχρεούται να το πράξει αυτό και εν προκειμένου επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι στην πράξη η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει πολλές τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεις. Από αυτές που ήδη θα δυνατόν να εκδώσει, η τελευταία, αν όχι η μόνη, είναι αυτή που αφορά τα σύνορα μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας και τους εσωτερικούς, τα εσωτερικά σύνορα και τους ελέγχους που έχουν επανεισαχθεί λόγω των δευτερογενών ε, μετακινήσεων που αποτελούσαν σοβαρούς κινδύνους για την ε, δημόσια τάξη και την ασφάλεια και που σήμερα είναι σημαντική πίεση για τα συστήματα των κρατών. Γιατί το λέω αυτό και γιατί επιμένω για αυτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής. Διότι βεβαίως σε σχέση με τα κρατη αυτό σημαίνει εκείνη τη διαδικασία διαβουλεύσεων για την ε, επαναφορά των ελέγχων στα ιστορικά σύνορα με συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί θα αποτελέσει έτσι ευκαιρία για πολιτικό διάλογο. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση της Επιτροπής για ε, έκδοση, για δυνατότητα η υποχρέωση έκδοσης γνωμοδότησης σημαίνει και διαδικασία διαβουλεύσεων και βέβαια συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά πάσα πιθανότητα. Επίσης υπάρχει μια ειδική νέα διαδικασία η οποία προβλέπεται στις περιπτώσεις όπου ο ίδιος σοβαρός κίνδυνος διαρκεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Και εδώ εισάγονται πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για να επιτραπεί αυτή η άρση ή η επαναφορα καλύτερα των ελέγχων, εκ των οποίων μία είναι ότι έχουν αναλυφθεί πρόσφορα εθνικά μέτρα από το κράτος μέλος μέσα στην επικρατεία του. Ένα κράτος υπεραδείγματι το οποίο ε, έχει ε, ανακηρύξει καθεστώς έκτακτης ανάγκης ή δυνάμει του εθνικού του δικαίου έχει ορίσει πως βρίσκεται σε ύψιστο επίπεδο κινδύνου, απειλής τρομοκρατικής επιθέσεως, μπορεί να γίνει δεκτό ότι είναι σε θέση να επαναφέρει, να διατηρήσει καλύτερα πάνω από τον ένα χρόνο τα ελέγχου στα ιστορικά σύνορα, εφόσον βεβαίως είναι συναφής με την απειλή. Σήμερα τέτοια περίπτωση τα κράτη-μέλη υποχρεώνται να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έξι μήνες πριν από την παράταση, πάλι γνωμοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ παράλληλα με το υφιστάμενο 29, άρθρο 29 και τη διαδικασία του, την τελευταία λέξη δεν την έχει το κράτος μέλος, επί τη βάση της γνωμοδότης Επιτροπής, το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για σύσταση προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να παρατείνει ή μη την διαρκεία της επαναφοράς των, των ελέγχων στα ιστορικά σύνορα. Αυτά, Πρόεδρε, εν ολίγης, αφορούν τις κύριες αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εφιστάμενο σύστημα της ρήτρας ασφάλισης. Επίσης, έχουμε σύσταση από την Επιτροπή ως συλλογικό όργανο, η οποία δίνει μια ερμηνεία των ισχύουσων διατάξεων υπό το πνεύμα των αλλαγών που προτείνονται από τις διατάξεις του κώδικα Σέγγεν των συνόρων. Άρα λοιπόν, εάν τα κράτη-μέλη τώρα κοινοποιούν την εισαγωγή ή παράταση των ελέγχων στα ιστορικά σύνορα, ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν και οι απαραίτητες επαφές με τα γειτονικά κράτη-μέλη, η συνεργασία, βεβαίως οι κοινοποιήσεις που γίνονται ε, σήμερα ή αύριο θα πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις του κώδικα σύνορων Σέγγεν. Και θα σας αποκαλύψω και το εξής, ότι λάβαμε από τη μια μέρα στην άλλη δύο κοινοποιήσει που θα πρέπει να έχει λάβει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μεταξύ, γιατί ταυτόχρονα θα πρέπει να μας έχουν κοινοποιηθεί, τόσο σε εσά, σε εμάς, όσο και στα κράτη-μέλη. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά αυτές τις κοινοποιήσει και προβαίνει στον αναστοχασμό των, της κατάλληλης συνέχειας που πρέπει να δοθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ντεκόιστερ. ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Κοέλιο, τον εισηγητή μα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και για τον ε, σαφέστατο τρόπο που μας τα είπε ο κύριος Κώστα. Όπως είπα χθε και στον Επίτροπο, σε γενικές γραμμές καλωσορίζουμε τις προτάσεις για μια στοχευμένη τροποποίηση του κώδικα Σέγγεν. Μάλιστα, οι πρόσφατες αυτές κρίσεις άσκησαν πίεση στον χώρο ελεύθερης ε, μετακίνησης ε, και τελικά καταλήξαμε σε επανεισαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε πολλά κρατημέλη και για μεγάλο διάστημα. Επίσης, ε, κατέστη σαφές ότι έπρεπε να αυξηθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, να αυξηθεί η δημοκρατική λογοδοσία και να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο σε περιπτώσεις εθνικής ασφαλείας. Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα την Σέγγεν από ελλείψεις, σεβόμενοι το δικαίωμα των κρατών μελών να προστατεύσουν τα σύνορά τους. Όμως, σήμερα πληροφορήθηκα ότι η Δανία, μία από τις δύο χώρες που ανέφερε ο κύριος Ντεκώστερ, είπε ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους ε, στα εσωτερικά σύνορα. Όπως ξέρετε, έχει φτάσει στο ανώτατο δυνατό χρονικό περιθώριο. Η Δανία επικαλέστηκε την τεράστια εισρωή ετούντων άσυλο. Ξαναλέω, τεράστια εισρωή ετούντων άσυλο και είπε τα εξής. 300.000 άτομα. 3 με 5 μηδενικά. 300.000 άτομα ελέγχθηκαν στα σύνορα μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου και για την ίδια περίοδο 263 άτομα ζήτησαν άσυλο στα σύνορα. Να υπενθυμίσω ότι επικαλέστηκαν τεράστια εισρωή ετούντων άσυλο. 263 άτομα. Δεν μιλάμε για 10% ή 5% ούτε για 1%. Μιλάμε για 0,1%. Τώρα ε, η περίπτωση της Ανίας λοιπόν φαίνεται ότι αφορά την ασφάλεια. Ποια στοιχεία έχουν δώσει για να το ε, δικαιολογήσουν αυτό. Εντυπωσιακά νούμερα, όπως αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, και η Κομισιόν με την στήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει παρουσιάσει ένα δικό χαρτί για να αναβιώσει την Σέγγεν. Σαφώς κάποια κράτη-μέλη λοιπόν έχουν διαφορετικό οδικό χάρτη και φοβάμαι ότι η Δανία είναι η πρώτη που ανοίγει τον δρόμο. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα κάνει η Κομισιόν για αυτή την κατάσταση. Θα επαναφέρουμε την Σέγγεν ή θα πεθάνει οριστικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και για την ανάλυση και τα παραδείγματα που μας δώσατε. Έχουμε ακόμη κάποιους βουλευτές που θέλουν το λόγο. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποθέτω ότι οι προτάσεις που βρίσκονται επί θα περάσουν από την κανονική διαδικασία. Θα προταθεί ένας εισηγητής, τροπολογίες, ε, ψηφοφορίες κτλ. Αυτό βεβαίως θα αργήσει. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η δυνατότητα της Γαλλίας για επιπλέον συνοριακούς ελέγχους ε, εξαντλείται στις 13 Νοεμβρίου υπό την υφιστάμενη νομοθεσία, ενώ οι δυνατότητες για Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Νορβηγία εξαντλούνται κάποια στιγμή το τέλος του Οκτωβρίου. Πώς τα συμβιβάζουμε αυτά. Υπάρχουν προτάσεις εδώ να επιτραπεί σε αυτές τις χώρες να έχουν συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, ενώ οι προτάσεις επιτάπητος σου επιτρέπουν να βάζεις ένα εξάμεινο και ένα εξάμεινο και ένα εξάμεινο αλλά εξαντλούνται προσεχώς υπό την τρέχουσα νομοθεσία. Και από ό,τι κατάλαβα από τις ε, αποκρίσει εδώ στο πακέτο, ένα κράτο μέλο μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικό πρόσχημα για να ξαναρχίσει τον έλεγχο στα σύνορα. Κάτι το οποίο υπονόησε και ο κύριο Κοέλιο με την Δανία, αλλά θεωρώ πω η Κομισιόν ουσιαστικά δίνει αυτό το επιχείρημα στα κράτη-μέλη. Αλλάξτε το πρόσχημα και ξαναρχίστε από το μηδέν. Έτσι είναι. Γιατί είναι πολύ ανησυχητικό. Γιατί αυτό δεν είναι επαναφορά της Σέγγεν που θα λειτουργεί όπως θέλουμε να λειτουργεί. Σας ευχαριστώ, Ζουντίθ, ο κύριος Κοράο και μετά η Μαρή Κριστίν Βερζιά. Σας ευχαριστώ. Προατήρουμε από αυτά που λένε και ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση για την ανθεώρηση του κώδικα συνόρων Σέγγεν είναι η απόδειξη, πιστεύω, του γεγονό ότι δεν έχουν το ίδιο βάρο, το ίδιο ειδικό βάρο όλα τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνε που ενοχλούν κάποια κράτη-μέλη πολύ εύκολα και γρήγορα προσαρμόζονται, θα έλεγα, παρότι παραβιάζονται κύριε αξίε Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η ελεύθερη διακίνηση στο χώρο Σέγγεν η αρχή της ελεγγύης ισχύει μόνο στα λόγια, ποτέ δεν μετατρέπεται σε έργα. Και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί κατάφορη απόδειξη αυτού του γεγονότος σήμερα. Στις 11 Νοεμβρίου εκπνέει τελική προθεσμία για ορισμένα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, για τη διατήρηση των, εσωτερικών, των ελέγχων στα ιστορικά σύνορα στον χώρο Σέγγεν. Μετά από αυτή δηλαδή θα μπορούσαν να διαφυλάξουν, να διατηρήσουν αυτού του ελέγχου χωρί να εκτεθούν σε κυρώσει. Και θα ήθελα προκειμένου να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ταχύτητα με την οποία έσπευσε να προσφέρει χείρα βοηθεία στα κράτη αυτά τα οποία ε, οθέτουν σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση του χώρου Σέγγεν. Και έτσι μπορούν να απαλλαγούν από οποιαδήποτε πίεση ή κυρώσεις. Φαίνεται ότι έτσι μπορεί σημαντικά να αυξηθεί η διάρκεια της παράτασης των ε, Ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για λόγου εσωτερική ασφάλεια και δημόσια τάξη, χωρί όμω καμιά εξωτερική αξιολόγηση. Μόνο το κράτο μέλο που επαναφέρει του ελέγχου έχει αυτή την αξιολόγηση και θα λέγω ότι το Νοέμβριο, όταν εκπνεύσει και η τελευταία δυνατή δυνατότητα παράταση, τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη δεν θα διστάσουν να διατηρήσουν του ελέγχου στα εσωτερικά του σύνορα στα εσωτερικά σύνορα. Το γεγονό ότι έχει κατευθεί πλέον αυτή η πρόταση αποτελεί επαρκή δικαιολογία για τα κράτη αυτά, αλλά και εγγύηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν πρόκειται να προβεί σε κάποια διαδικασία επί παραβάση ει βάρο του. Επίση, η διασύνδεση μεταξύ της απειλής ε, για την ασφάλεια και τη μετανάστευση στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σημειώνουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο το ότι οι δευτερογενείς κινήσεις θεωρούνται λόγος κίνδυνης και ότι, κινδύνουν και ότι οι μετανάστες θεωρούνται απειλή τρομοκρατική. Η τροποποίηση μιας κατάστασης τέτοιας όπως αυτή της απειλής για την εσωτερική ασφάλεια ή δημόσια τάξη δεν μπορεί να μπαίνει στο πλαίσιο Σέγγεν όταν δεν υπάρχει ενίσχυση τη δυνατότητα ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα μέσω της περιοδικής αναθεώρησης Σέγγεν γιατί μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν ε, καταχρήσεις που έχουν να κάνουν με τα κράτη της πρώτης άφηξη. Τα εξωτερικά σύνορα δηλαδή έχουν μετατραπεί πλέον και τα κράτη που έχουν τα, τα εξωτερικά σύνορα μετατρέπονται σε στρατόπεδα υποδοχής προσφύγων ενώ δεν προχωρούμε καθόλου σε θέματα μετανάστευση. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακριβώς ορισμένα κράτη να παραμείνουν ω καταπλησμοί προσφύγων ε, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοράου. Μαρή Κριστίν. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπάμαι αλλά έχασα ένα κομμάτι της ε, παρουσίασης γιατί ήμουν σε μια άλλη συνεδρίαση. Ήθελα να επαναλάβω αυτό που έχω ήδη πει σε σχέση με την ανησυχία μου για τα ε, γαλλοϊταλικά σύνορα Για να θυμίσω ότι η Γαλλία δεν βασίζεται στα ίδια άρθρα όταν ζητά την επαναφορά των συνόρων. Στηρίζεται στο 25, αλλά όχι και στο 29, αλλά στο 27 αν κατάλαβα καλά τις εξηγήσει της Κομισιόν, αυτό της δίνει πολύ μεγαλύτερο περιθώριο λιγμού και δυσκολία ελέγχου, πολύ μεγαλύτερη επίσης για την Επιτροπή αλλά με ανησυχεί πάρα πολύ και το ξαναλέω για τα όσα συμβαίνουν στα γαλλικά σύνορα. Γιατί η Γαλλία χρησιμοποιεί την τρομοκρατία για να, μάλλον επικαλείται την τρομοκρατία για να επαναφέρει τα σύνορα, αλλά στην ουσία κάνει έλεγχο των μεταναστών και για λόγους ε, έκδηλη συμπαράσταση στην Ιταλία, γιατί στην Γαλλία δεν υπήρξε αύξηση μεγάλη των μεταναστών, αντίθετα με το τι συνέβη στην υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως στην Γερμανία. Όσον αφορά λοιπόν τα γαλλογιταλικά σύνορα, υπήρξαν 30.000 αρνήσεις εισόδου στην επικράτεια της Γαλλίας. 30.000. Ξέρουμε ε, ότι από αυτές τις 30.000 ε, επανειλημμένως τους απαγορεύθηκε η είσοδος αλλά στα χάλο-ιταλικά σύνορα, μόνο για το Ισάλπ Μαριτίμ ε, και την Ιταλία, έχουμε το 70% των απαγορεύσεων εισόδου στα σύνορα της Γαλλίας. Και, εδώ μεταξύ, 700 με 800 αιτήσει για άσυλο κατατέθηκαν στην ίδια αυτή, στον ίδιο αυτό νομό για το 2016. Υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία, λοιπόν. Να πω λοιπόν στην κυρία Σαργεντίνη ότι η Γαλλία ήδη ζήτησε την παράταση της ε, ισχύω των συνόρων δεν έχω... μέχρι τις 30 Απριλίου 2018. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω δεν έχω ακριβώς το, τώρα το αίτημα ε, σε τι στηρίζεται η Γαλλία για να συνεχίσει να κάνει συστηματικούς ελέγχους στα σύνορα και λέω ότι κάνει ελέγχους ε, φάσιες, δηλαδή ε, τεράστιες διακρίσεις. κατάλαβα καλά αυτό που είπε η Επιτροπή. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθείτε να φτιάξετε μια δέσμη μέτρων ώστε να μην υπάρχουν δύο πηλαίων δυνατότητε, αλλά μόνο μία δυνατότητα αίτηση τη επαναφορά των συνόρων. Για να μην υπάρχει αυτή η, η διαφορά ανάμεσα στο 27 και στο 29. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να επανέλθω στον κύριο Ντεκόιστερ, ώστε να του δώσω το λόγο και να απαντήσει σε όλε αυτέ τι ερωτήσει. Η κυρία Σαργεντίνη αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική απάντηση. Τι κάνουμε εμείς ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Οπότε θα ζητήσω τον κύριο Ντεκόιστερ να απαντήσει για την Κομισιόν, αλλά ο κύριος Κοέλιο που είναι ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας της ΛΥΜΠΕ για το ΣΕΝΚΙΝ για την ασφάλεια θα μπορούσε να μας πει ακόμα κάποια πράγματα για το πού κινούνται οι προσπάθειες για τη δική μας προσέγγιση. Έχουμε, έχουμε και συνάντηση των συντονιστών στις 23 ε, Αλλά σε αυτό θα επανέλθω αφού θα ακούσουμε τον κύριο Τεκόιστερ. παρατηρήσεις λοιπόν που μας ανησυχούν. Κύριε Δεκόιστερ λοιπόν, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις παρατηρήσεις. Thank you, Mr. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω γενικά σε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Ε, προκλητική ερώτηση που έγινε από τον κύριο Κουαλιό. Εδώ αν η Κομισιόν θέλει να ξαναλειτουργήσει η Σέγγεν ή αν την έχει εγκαταλείψει. Από όλα τα έγγραφα, την πολιτική επικοινωνία, τις νομοθετικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί προσφάτως και αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, πρέπει να είναι σαφές ότι η Κομισιόν βεβαίως θέλει να επανέλθει η Σέγγεν έχει υποβάλει όλες τις απαραίτητες προτάσεις για να γίνει αυτό. Για τον σκοπό αυτό, λοιπόν. Αλλά προφανώς δεν αρκούν αυτά μέχρι στιγμής. Αλλά είμαστε σαφείς. Η Κομισιόν, το έχει πει και ο πρόεδρος Γιούνκερ, η Σέγγεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα για τους πολίτες της. Δεν πρέπει να χάσουμε τα ωφέλη της Σέγγεν για τους πολίτες. Τούτου λεχθέντος. Αφετέρου υπάρχουν πράγματι προκλήσεις στην πλευρά της ασφαλείας που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ας είμαστε όμως αφείς. Εάν αποφάσιζε μόνο η Κομισιόν, θα επαναφέραμε την Σέγγεν χτες και όχι αύριο. Δεύτερον, κάποιος είπε ότι η Κομισιόν δίνει πρόσχημα στα κράτη-μέλη για να παρατείνουν τους ελέγχους και τους λέμε να διαλέξουν άλλους λόγους. Επ' αυτού, κύριε Πρόεδρε Κομισιόν, καθόλου δεν κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι σαφές και σύνηθες νομικό δόγμα ότι αν επαναφέρεις ε, συνοριακούς ελέγχους για διαφορετικό λόγο κάθε φορά ξαναρχίζει το χρονόμετρο από την αρχή. Εάν επανέλθουν π.χ. Ε, σύλλογοι για ε, έλεγχοι για χουλιγανισμό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό μπορεί να γίνει. Αν ένα μήνα μετά την άρση των εσωτερικών ελέγχων επαναφέρει στους συνοριακούς ελέγχους γιατί έχει υπάρξει τρομερή ε, τρομοκρατική επίθεση ε, το δίμηνο που προηγήθηκε δεν μετράει για το εξάμηνο το maximum αυτή είναι η παραδοσιακή ερμηνεία των διατάξεων που κανείς δεν έχει ποτέ αμφισβητήσει κάτι άλλο είναι ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να είναι δημιουργικά όσον αφορά τους λόγους αυτούς και γι' αυτό ακριβώς σήμερα δεν είμαι σε θέση να πω ποια θα είναι Κομισιόν ε, η αντίδραση Κομισιόν στις νέες ε, κοινοποίησεις. Ε, τις λαμβάνουμε κυριολεκτικά το προηγούμενο βράδυ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν και τυπικότητες στην ειδοποίηση αυτή. Ξέρετε, διατυπώσεις η Κομισιόν επιμένει, παραδείγματος χάρη, να έχει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ε, για το μήπως επαρκούν ε, άλλα μέτρα, παραδείγματος χάρη, να αστυνομική έλεγχη εντός της επικράτειας, για να μην φτάσουμε στο μέτρο της εισαγωγής συνοριακών ελέγχων. Ε, αυτά τα πρίσματα ε, εξετάζουμε τις κοινοποίησεις και μετά το Σώμα των Επιτρόπων θα αποφασίσει τι συνέχεια θα δοθεί. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να σας απαντήσω σε αυτήν την φάση για τις ερωτήσεις και τα σχόλια που έγιναν. Και είμαι σίγουρος ότι στο προσεχές μέλλον θα υπάρξει μια πολιτική συζήτηση για το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεκόιστερ για την απάντηση. Είναι ε, ξόχος πολιτικό το ζήτημα και σας ευχαριστώ και για την ειλικρίνεια στην απάντησή σας. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε κάτι στη γραμμή που πρότεινε η κυρία Σαρτζαντίνη. Δηλαδή, πού στεκόμαστε εμείς σε σχέση με αυτά τα πολιτικά και τεχνικά ζητήματα της Λοιπόν, το νόημα της σημερινή συζήτηση, πέρα από το να ξανακούσουμε την Κομισιόν, είναι να διαμορφώσουμε μια απάντηση. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στα λίγα λεπτά που μας απομένουν να είναι να μας πει ο κύριος Κοέλιο το τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει τώρα το Κοινοβουλίο. Αυτό το οποίο θα πρότεινα εγώ ως κατεύθυνση είναι να ορίσουμε εισηγητή στην συνεδρίαση των συντονιστών του Οκτωβρίου, αλλά δεν θέλω τώρα αυτό να εμπλέξει το πρόγραμμα της ομάδας εργασίας. Οπότε αν μπορείτε να δείτε τι άποψη έχει η ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Πείτε μας λοιπόν την άποψή σας για να αντιδράσουμε, αλλά πρέπει να έχουμε έτοιμες αυτές τις επιλογές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να πω στους συναδέλφους το εξής. Αντιλαμβάνομαι την πρόταση της Κομισιόν γιατί την πρώτη φορά ετέθη το ζήτημα από την κυρία Βερζιά σε συνεδρία σύσκευων εισηγητών για το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού κίδεου όσον αφορά την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και κατά την άποψή μου η πρόταση της Κομισιόν προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτό το κενό. Αλλά πίσω από αυτό ανησυχούμε και υπάρχουν λόγοι ανησυχίας γιατί δεν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις καταστάσεις που θα έχουμε εσωτερικούς ελέγχους ε, στα σύνορα. Ε, αυτό θέλουμε ακριβώς ε, να ακολουθήσουμε την ιδέα που πρότεινε η Κομισιόν. Τι κάνουμε τώρα στην ομάδα εργασίας. Είχαμε πολλές συναντήσεις με καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιες από αυτές ήταν και κλεισμένων των θυρών. Λάβαμε ενημέρωση για το πρόβλημα, οπότε έχουμε μια καλή εικόνα του τι συμβαίνει και ξεκινάμε ήδη μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, ζητήσαμε την άδεια για την κατάσταση της Σέγγεν. Θα εγκριθεί αυτή η έκθεση και θα γίνει αυτή η συζήτηση στην συνεδρίαση στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια όταν φτάσει η στιγμή. Πρέπει να συνεδριάσει η ομάδα μόνο για τα εσωτερικά σύνορα στην επόμενη συνεδρίασή μας και τον Δεκέμβριο έχουμε μια συνεδρίαση για την Σέγγεν και πιθανώς οι συντονιστές θα πρέπει να σκεφτούν το πεδίο εφαρμογή. Είχαμε ε, σκεφτεί κάποιο στενότερο πεδίο εφαρμογή. Ε, δηλαδή η ακρόαση να είναι εσωτερική ακρόαση. Αλλά με βάση τα τελευταία γεγονότα θα έπρεπε να προσκαλέσουμε και τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό βεβαίως θα το βρείτε εσείς με τους συντονιστές. Εμείς μπορούμε να σας πούμε την άποψή μας. Αλλά μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, μία συζήτηση στο Κοινοβούλιο και μία συζήτηση για την κατάσταση της Σέγγεν, το Κοινοβούλιο θα σχηματίσει άποψη για το τι συμβαίνει στην Σέγγεν και αυτό μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας βοηθήσατε νομίζω αρκετά. Η ιδέα για την ακρόαση είναι πολύ καλή. Θα την εξετάσουν οι συντονιστές της 23. Θα μας πείτε βεβαίως και άλλα εσείς πριν γίνει αυτό. Μπορεί και να έρθετε και σε αυτήν την συνεδρίαση. δεδομένο του εύρους και της ευαισθησίας του Δήμου. Μ' αρέσει η ιδέα των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων ή της διάστασης των κρατών μελών για την ειλικρίνεια της απάντησης ε, γιατί, για, για να είμαστε ειλικρινείς βέβαια το θέμα είναι και των κρατών μελών, αλλά πρέπει να προσέξουμε. να μην έχουμε τις ε, συνήθεις, ε, τυπικές απαντήσεις και την συνήθη προσέγγιση. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και καιρό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ευέλικτοι. Δεν έχει νόημα να κάνουμε καμία συνεδρίαση η οποία θα είναι μακροσκελής και δεν θα επιτύχει το στόχο της. Ας δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε στις 23. Να δούμε λοιπόν και με τους συντονιστές και με τα μέλη της ομάδας εργασίας. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ευχαριστούμε την Κομισιόν, ευχαριστούμε κύριε Ντεκόιστερ, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσία σας, για το ένα θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.